Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε τη συνεδρίαση. Είναι κοινή συνεδρίαση μεταξύ δύο επιτροπών, ΑΦΚΟ και Γιούρι, ή Γιούρι και ΑΦΚΟ. Και αρχίζουμε αμέσως με την πληροφορία ότι καλέσαμε τον Κίφερ Χόφσταντ που τελείωσε τις διαπραγματεύσεις για την καλύτερη νομοθεσία και θα θέλαμε να μας κάνει την παρουσίαση προς τις δύο επιτροπές των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων αυτών και μετά θα μπορέσουμε να θέσουμε ερωτήματα και να λάβουμε και απαντήσεις. Ένας από τη Γιούρη, ένας από την Αύκο κάθε φορά. Γι' αυτό να το δηλώνετε εκ των προτέρων για να κάνουμε την εναλλαγή. Um, uh, uh, just maybe,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 Thank, thank you very much. So first of all, thank you very much uh, to uh, the chair of AFCO and the chair of uh, URI uh, to have this. Uh, uh, που διοργάνωσαν αυτή την κοινή συνεδρίαση προκειμένου να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για την καλύτερη νομοθέτηση στη Διοργανική Συμφωνία για την καλύτερη νομοθέτηση Όπω γνωρίζετε την περασμένη Τρίτη 8 Δεκεμβρίου ε, διεξήχθη τελική συνεδρίαση με συμμετοχή της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Στόχος ήταν να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις. Η συνεδρίαση πήγε καλά και έχουμε μια προσωρινή συμφωνία η οποία επιβεβαιώθηκε από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έλαβε τη θετική γνώμη της διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα το πρωί. Ε, σύμφωνα με την επίσημη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η διαδικασία είναι διαφορετική από την, αυτήν του Συμβουλίου ε, εμείς ε, δεν έχουμε μόνο ένα συλλογικό όργανο όπως η Κομισιόν, ούτε μόνο μια συνεδρίαση υπουργών που βρίσκονται από καιρούς καιρών όπως το Συμβούλιο. Εμείς εδώ έχουμε επιτροπές, είμαστε οργανωμένοι σε επιτροπές που προετοιμάζουν μια γνωμοδότηση η οποία τελικά ψηφίζεται στην Όλο μέλε και πράγματι αυτό θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. έστειλα στις υπηρεσίες της ΑΦΚΟ ε, το, και της Γιούρη το κείμενο, το τελικό κείμενο καθώς επίσης και ένα σημείωμα μ, επεξηγηματικό ανακεφάλαιο του περιεχομένου της συμφωνίας. Οπότε αυτό που απομένει να κάνω σήμερα δεν είναι προφανώς να σας αναγνώσω το κείμενο της συμφωνίας, κάτι που θα ήταν βαρετό. Μπορώ όμως να σας κάνω μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων. Με άλλα λόγια, ποια είναι τα καινούρια στοιχεία, ποια είναι τα επιτεύγματα, τι το καινοτόμο έχει αυτή η διοργανική ε, συμφωνία ποια είναι αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν υφίσταντο στην προηγούμενη συμφωνία του 2003. Και δεν μιλώ για την συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου του 2010, γιατί εκείνη η συμφωνία εξακολουθεί να είναι ενισχύ. Υπάρχει μια ε, δήλωση των δύο οργάνων, Κομισιόν και Κοινοβουλίου, ότι αυτή η συμφωνία εξακολουθεί να ισχύει. Η συμφωνία πλαίσιο. Ε, τώρα πλέον έχουμε τρεις, τρία όργανα ε, και γιατί, γιατί το Συμβούλιο ζήλεψε λιγάκι τα τελευταία χρόνια επειδή υπήρχε μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Κομισιών Κοινοβουλίου και για πρώτη φορά ζήτησε το Συμβούλιο να γίνει μια τριμερής συμφωνία και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη κατά την άποψή μου. Γιατί? Γιατί κινούμαστε προς μια κατεύθυνση όπου η Κομισιόν ε, θεωρείται όλο και περισσότερο ως εκτελεστικό όργανο, δεν θα έλεγα κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά γιατί δεν είναι κυβέρνηση, ε, εκτελεστικό όργανο με δικαίωμα πρωτοβουλίας, κάτι το οποίο είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, και δύο νομοθετικά όργανα, Παρόλο ότι το Συμβούλιο έχει και κάποιες εκτελεστικές αρμοδιότητες που ενδεχομένω ε, θα εξαφανιστούν τα επόμενα χρόνια με τις επόμενες ε, συνθήκε που ενδεχομένω θα υπογραφούν. Το Συμβούλιο πάντω, ήθελε να διαπραγματευτεί με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο πέραν και παράλληλα τις ε, συμφωνίας πλαίσιο του 2010, μία διοργανική συμφωνία μεταξύ των τριών λοιπόν θεσμικών οργάνων, ε, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει την δομή αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίγωνο. Ένα εκτελεστικό όργανο, την Κομισιόν και δύο νομοθετικά όργανα, ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που αντιπροσωπεύουν τις κυβερνήσεις και τα, τους λαούς αντίστοιχα. Αυτό είναι κάτι το οποίο τόσο η ΑΦΚΟ όσο και η Γιούρ και γενικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιζητούσαμε εδώ και πολύ καιρό. Ε, μπορώ να πω μάλιστα ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ε, δεν είδα και μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Πιο πολύ με την Κομισιόν θα έλεγα, ε, παρά με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ήταν ε, από την πλευρά των διακριτητών συγκεκριμένων πραγμάτων, ζητούσαν από την Κομισιόν. Τώρα, ποια είναι τα καινούργια στοιχεία. Οκτώ χαρακτηριστικά μπορώ να ξεχωρίσω. Οκτώ νέα σημεία στα οποία έχουμε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις σε σχέση με το, το τι ισχύει σήμερα. Για πρώτη φορά τα τρία θεσμικά όργανα αναλαμβάνουν ευθύνε για, το ετήσιο και το για τον ετήσιο και πολιετή προγραμματισμό του, του έργου. Το άρθρο 17 της ε, συνθήκης ε, το προβλέπει. Συμφωνήσαμε στην αρχή κάθε νομοθετικής περίοδου τα τρία θεσμικά όργανα να συμφωνούν για ένα, για ένα κατάλογο προτεραιοτήτων ε, ε, πολιετούς διάρκειας. Και επιπλέον κάθε χρόνο, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα της εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να εγκρίνουμε μια κοινή δήλωση για τις κοινέ νομοθετικές προτεραιότητες των τριών οργάνων. Οπότε θα έχουμε προτεραιότητε για όλη την νομοθετική περίοδο, τα πέντε χρόνια δηλαδή, και μετά θα έχουμε προτεραιότητε κάθε χρόνο. Μία πλέον παρατήρηση. Το γεγονό ότι το κάνουμε αυτό τόσο ρητά πλέον σημαίνει ότι στην ενδιάμεση αξιολόγηση του χρηματοδοτικού πλαισίου, δημοσιονομικού πλαισίου, ε, θα πρέπει να δούμε τις προθεσμίες. Γιατί δεν είναι δυνατόν το ε, δημοσιονομικό πλαίσιο να έχει περίοδο 7 ετών και η νομοθετική περίοδος 5 ετών διάρκεια. Οπότε αυτό θα πρέπει να το δούμε στην ενδιάμεση αξιολόγηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ε, θα δίνει τη γνώμη του για την απόσυρση προτάσεων πλευρά κομισιών, για την απλοποίηση προτάσεων πλευρά κομισιών και επίση θα έχουμε και μια διαδικασία διότι αφορά την παρακολούθηση ε, των ετοιμάτων ε, νομοθετική πρωτοβουλία από, από ένα από τα δύο όργανα. Για παράδειγμα, όταν έχουμε μια εκθέσει ε, ε, πρωτοβουλία η ίδια πρωτοβουλία νομοθέτηση, η Κομισιόν θα πρέπει να δίνει μια συνέχεια η οποία θα παρακολουθείται με συγκεκριμένο τρόπο. Έχουμε λοιπόν ε, προτερότητες πολιετής, μονοετής και θα δίνουμε τη γνώμη μας για τις αποσύρσεις απλοποίησης και, τα αιτήματα του, και τη συνέχεια που δίνεται στα αιτήματα νομοθετικής δράσης. Δεύτερον, διευκρινίζουμε πλέον την ε, χρήση των ε, μελετών αξιολόγηση αντικτύπου. Δεν ήταν εύκολο από πλευρά μα. Γιατί ε, ούτε εντό του κοινοβουλίου είχαμε ενιαία άποψη, κοινή άποψη. Ενδεχομένως και εξετάζοντας το αποτέλεσμα της συμφωνίας μπορεί να μην έχουμε ε, μια ομοφωνία σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του δηλαδή. Πάντως το θέμα ήταν να, ε, να ξεκαθαρίσουμε το θέμα της ε, αξιολόγησης αντικτύπου. Ε, έχουμε ξεκαθαρίσει το ποιου τομεί θα καλύπτει, οικονομικού, περιβαλλοντικού, ε, κοινωνικές, κοινωνικό αντίκτυπο, ε, ανταγωνιστικότητα τη οικονομία, ε, διοικητικό άχθο, ε, ε, το κόστος της μη Ευρώπης, το ψηφιακό ε, και το χωρικό. Δηλαδή αν επηρεάζει περισσότερο το ένα τμήμα της Ευρώπης και λιγότερο κάποιο άλλο και βέβαια το πώς επηρεάζει της οικονομική η κάθε νομοθετική πράξη. Η Κομισιόν αναλαμβάνει αυτή την αξιολόγηση, αλλά εξασφαλίσαμε σύμφωνα με την διαπραγματευτική εντολή που δέχθηκα από το Κοινοβούλιο, εξασφαλίσαμε ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να κάνουν το, τη δική του αξιολόγηση ε, για τις δικές τους τροπολογίες αν το θεωρούν απαραίτητο. Από πλευρά της Κομισιόν θα χρησιμοποιήσουν ένα ανεξάρτητο ρυθμιστικό συμβούλιο Αξιολόγηση. έτσι ώστε οι προτάσει του να αξιολογούνται με αντικειμενικό τρόπο και επειδή αυτό το Συμβούλιο θα είναι εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησα πριν το τέλος των διαπραγματεύσεων να ενημερωνόμαστε για το πώς θα εργαστεί θα εργάζεται αυτό το Συμβούλιο. Διότι το αναφέρουμε στη Συμφωνία. Άρα λοιπόν λογικό είναι να γνωρίζουμε πώς το Συμβούλιο, ε, Κανονιστικό Συμβούλιο Αξιολόγησης θα εργάζεται. Και λάβαμε από τον κύριο Τίμερμανς μια τρισέλιδη εξέταση, λεπτομερέστατη εξήγηση, ε, για το πώς θα λειτουργεί το Συμβούλιο, έγγραφο το οποίο μάλιστα σας έστειλα, έστειλα στις δύο επιτροπές και στο, στη διάσκεψη των πρόεδρων γιατί αυτή η επιστολή ε, που θα πρέπει να προσαρθεί και στη δική μας ε, έκθεση, στη δική σας έκθεση, ε, περιλαμβάνει, λέω, λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργεί αυτό το Συμβούλιο Αξιολόγησης Αντικτύπου ε, των Προτάσεων της Κομισιόν. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Διευκρίνηση λοιπόν της ε, χρήσης ε, του εργαλείου της αξιολόγησης αντικτύπου. Χωρίς να υποσκάπτουμε τις νομοθετικές εξουσίες των δύο οργάνων, διευκρινίζουμε το πώς θα λειτουργήσει ε, αυτός ο θεσμός και το πώς θα εξασφαλιστεί η αμεροληψία και η αντικειμενικότητά του. Τρίτο στοιχείο. Το θέμα της αλλαγής της νομικής ε, βάσης, πράγμα το οποίο εμφανίζεται αρκετά συχνά. Γνωρίζετε ότι στο μέσο της νομοθετικής διαδικασίας, μερικές φορές και στο τέλος, στο τέλος, στο τελευταίο, στην τελευταία συνεδρία του τριμερούς διαλόγου, κατά τύχη μερικές φορές δήθεν, το Συμβούλιο αλλάζει τη νομική βάση ε, και αποφεύγει την, με αυτόν τον τρόπο την ε, συνομοθεσία ε, κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά να προσφύγουμε στο ε, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πλέον, το Συμβούλιο πλέον όταν θέλει να σκέφτεται να αλλάξει την νομική βάση θα πρέπει να συγκαλεί τριμερή συνάντηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να σταματήσουμε την αλλαγή, έτσι αυτή είναι μια απόφαση του Συμβουλίου, αλλά έχει πλέον υποχρέωση το Συμβούλιο να συγκαλεί ε, συνάντηση των τριών σωμάτων σε περίπτωση που σκέφτεται να αλλάξει την νομική βάση ε, κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Και η Κομισιόν έχει υποχρέωση να υπερασπιστεί της αρχικής της επιλογής. Ε, επιλογή της νομικής ε, βάσης ε, άλλες φορές ε, προκύπτει από την ίδια τη συνθήκη και άλλες φορές από την ερμηνεία που δίδεται σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου και θα πρέπει η Κομισιόν είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο τρόπο να υπερασπίζεται την αρχική επιλογή που έχει κάνει. Αυτό λοιπόν είναι το τρίτο στοιχείο στην περίπτωση που το Συμβούλιο έχει σκοπό να αλλάξει νομική βάση. Τέταρτο νέο στοιχείο για τις κατεξιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Δεν θέλουμε οι, ε, δεν μας αρέσουν ε, οι εφαρμοστικές πράξεις, ε, μας ενδιαφέρουν περισσότερο η κατεξιοδότηση πράξης. Και επειδή τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο δεν εμπλέκονται στις κατεξουδότηση πράξεις ε, ενδιαφέρονται περισσότερο να εκδίδονται ε, εφαρμοστικές πράξεις. Οπότε εκεί είχαμε μια μικρή σύγκρουση συμφερόντων. Για να διευκολύνουμε τη χρήση των κατεξουδότηση πράξεων συμφωνήσαμε ότι ε, στην προετοιμασία αυτών των πράξεων θα ερωτώνται, ε, θα δίνουν ε, τη γνώμη τους και τις συμβουλές τους εθνικοί εμπειρογνώμονες και το κοινοβούλιο θα έχει την ίδια πρόσβαση σε αυτές τις συνεδριάσεις που θα έχουν και οι εθνικοί εμπειρογνώμονες καθώς επίσης και στα έγγραφα θα έχει την ίδια πρόσβαση που θα έχουν τα κράτη-μέλη. Οπότε θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο θέμα του πότε θα χρησιμοποιούμε το ένα τύπο πράξεων και το πότε θα χρησιμοποιούμε τον άλλο τύπο πράξεων, ε, έχουμε μία ε, ρήτρα ε, στη συμφωνία η οποία θα λέει ότι μόλις θα τεθεί σε, συμφω... ισχύ ε, η συμφωνία θα ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση διαπραγμάτευση για τον, τη διευκρίνηση των κανόνων για το πότε θα ο, χρησιμοποιούνται οι, κατεξιοδότηση πράξεις και πότε ε, οι εφαρμοστικές πράξεις. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί θα προκύψουν διαφωνίες για το τι είδους πράξη θα χρησιμοποιείται κάθε φορά οπότε χρειαζόμαστε απαραίτητα αυτά τα κριτήρια. Ε, δεν έχουν προβλεφθεί συμφωνία, θα ξεκινήσει η διαπραγματευσή τους μόλις τεθεί σε ισχύ συμφωνία. Ε, αυτή τη στιγμή η διαδικασία διευκολύνει τη χρήση των εκτελεστικών πράξεων ε, η συμφωνία όμως, η διοργανική συμφωνία την οποία, στην οποία καταλήξαμε θα ε, ευνοεί περισσότερο τις κατεξοδότηση πράξεις κάτι που θα μειώνει τη σημασία του ρόλου του Συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά η διαπραγμάτευση ε, για τα κριτήρια χρήση της μια, του ενός του άλλου τύπου θα ξεκινήσει μετά την θέση της συμφωνίας. Πέμπτο καινοτόμο στοιχείο Βελτιώσαμε τη διαφάνεια σε ένα αριθμό σοβαρών σημείων. Υπάρχει ένας αριθμός διατάξεων και πρόνοιων που ευνοούν τη διαφάνεια. Δεν σας τις αναφέρω όλες. Για παράδειγμα όμως ε, θα έχουμε ένα ε, κατάλογο, ένα μητρό ε, κατεξιδότηση πράξεων που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Θα δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του 2017 θα έχουμε μια κοινή βάση δεδομένων νομοθετικών φακέλων, οπότε θα παρακολουθούμε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο κάθε φάκελος ηλεκτρονικά. Προβλέπετε μια καλύτερη διαφάνεια στην όλη διαδικασία συμπεριλαμβανομένης και της απαραίτητης, του απαραίτητου επίπεδου διαφάνειας των, των τριμερών διαλόγων. Και όταν λέω απαραίτητο, είναι προφανές τι σημαίνει αυτό. Το, ο τριμερής διάλογος δεν είναι κλασικό κομμάτι της ε, νομοθετικής διαδικασίας. Ε, δεν είναι δυνατόν τριμερής διάλογος να γίνεται στην Grand Place των Βρυξελών και να είναι τελείως ανοιχτός. Ε, αλλά χρειαζόμαστε ένα ελάχιστο επίπεδο διαφάνειας για, τον, για τους τριμερείς διαλόγους. Θα το συζητήσουμε βέβαια στο μέλλον ποιο είναι αυτό το κατάλληλο επίπεδο διαφάνειας, ε, αλλά ήδη συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία. Οπότε έτσι ικανοποιούμε το αίτημα του Ombudsman, ε, του διαμεσολαβητή του Κοινοβουλίου, ε, που έστειλε μάλλον μια επιστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ε, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη διαφάνεια στους τριμερείς διαλόγους. Ικανοποιούμε λοιπόν και το δικό του αίτημα. Έκτο στοιχείο και καινοτομία. δεν είναι εύκολο βέβαια. Είναι η αρχή τις ίσης ε, θέσεις Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όταν συνομοθετούν. Δηλαδή, εμείς που είμαστε δημοκρατικό όργανο, ε, συνεδριάζουμε δημόσια, είμαστε ανοιχτά, μπορεί να έρθει όποιος θέλει το Συμβούλιο, στην Επιτροπή σας, στη Γιούρη, στην ΑΦΚΟ ε, και στην Ολομέλεια. Το αντίστροφο είναι διαφορετικό. Κάποιος ρωτάει γιατί. Ε, ο Γιολάινεν. Δεν ξέρω γιατί γιο, όλα έτσι είναι τα πράγματα, έτσι έχουν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ανοίξουμε τη ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Για το κοινοβούλιο ήταν πάντα κλειστή, ανέκαθεν αυτή η πόρτα, θεός φράγιστη. Υπάρχουν διάφορες πρακτικές που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις επαφές και το συντονισμό και ε, θα έχουμε τακτικά ε, τα δύο θεσμικά όργανα άτυπες ανταλλαγές απόψεων και εγγράφων φυσικά άτυπα, το ξέρω είναι αυτά, αλλά είναι τουλάχιστον η αρχή μιας νέας διαδικασίας. Μάλλον δεν θα είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα διαπραγματευτεί τη νέα συμφωνία, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, αλλά έχει ανοίξει μια χαραμάδα και είναι γεγονός η άτυπη ανταλλαγή απόψεων συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων. Και επίση έχουμε προβλέψει και κάτι διαφορετικό. Πρόκειται για την καλύτερη νομοθεσία, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με τι διεθνεί συμφωνίε, αλλά έχουμε και μια ρήτρα ραντεβού για την αρχή διαπραγματεύσεων για μια διοργανική συμφωνία έξι μήνε μετά τη θέση σε ισχύ της ε, παρούσης για ε, τα θέματα πλέον διεθνών συμφωνιών. Γιατί αρχή ε, βρίσκεται στη συνθήκη, το έχουμε ε, εγκρίνει από τη της τηλεφώνας και μετά ως κοινοβούλιο έχουμε νέα αρμοδιότητα, αλλά ουδέποτε, ουδέποτε ε, είχαμε διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σημαίνει αυτό στην πρακτική και τα διάφορα στάδια των διαπραγματεύσεων. Εγώ έλεγα απορρίψαμε την άκτα, απορρίψαμε το SWIFT, μπορεί και άλλες ενδεχομένως στο μέλλον διεθνείς συμφωνίες, αλλά αυτό δεν μας βοηθάει να προχωρήσουμε παρακάτω και δεν βοηθάει και το Συμβούλιο. Πρέπει να τα βρούμε, πρέπει να τα βρίσκουμε. Γι' αυτό προβλέπεται αυτή η ρήτρα για το πότε θα ξεκινήσει. Δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ε, ε, πάντως χρειάζεται διοργανική ε, συμφωνία για τις διεθνείς συμφωνίες, επαναλαμβάνω, και θα αρχίσει αυτή έξι μήνες μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσης. Έβδομο σημαντικό νέο στοιχείο. Και τώρα έρχομαι σε κάτι που για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Α, αυτό που λέμε gold plating, λέει η κυρία Χιούβνε. Ναι, ναι, αυτό δεν είναι ότι μου αρέσει εμένα το χρυσάφι ή το επιχρήσωμα. Εντάξει, σε ποιον δεν αρέσει ο χρυσός, αλλά επειδή 9 χρόνια το έκανα ε, αυτό το gold plating που είναι η εθνική νομοθεσία επί της κοινοτικής. Αφού το έκανα λοιπόν εγώ ε, ως πρωθυπουργός, ρωτήστε στο Βέλγιο, γιατί είμαστε ειδικοί. Ήταν λοιπόν ε, μεγάλη μάχη αυτή που δόθηκε με το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για το πώς περιορίζεται η αυτονομία των κρατών μελών στη διαδικασία λήψεων αποφάσεων. Δεν περιορίζεται. Δεν τους λέμε ότι δεν μπορείτε να έχετε εθνικέ ρυθμίσεις επιπλέον, αλλά στο εξή αυτό θα πρέπει να είναι πάρα πολύ πώς να το περιορισμένο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει λόγο ποια είναι η μεταφορά της οδηγία και ποια είναι η εθνική νομοθεσία που έρχεται να βαρύνει ακόμα παραπάνω την οδηγία αυτή που μεταφέρεται. Γιατί μέχρι τώρα τι συμβαίνει. Ευρώπη σου λένε, η Ευρώπη μας τα έχει επιβάλει όλα αυτά και είναι υπεύθυνη ή φταίει για την υπερβολική ρύθμιση, για την υπερβολική γραφειοκρατία. Ενώ στην ουσία τι συμβαίνει. 50-50, για να μην πω ότι καμιά φορά και παραπάνω είναι ένα κεφάλαιο που έχει έρθει να προσθεθεί σε εθνικό επίπεδο στις διαπραγματεύσεις. Άρα θα ελέγχεται αυτό και θα περιγράφεται και θα εξετάζεται ξεχωριστά έτσι ώστε να μπορούν οι πάντες να ξέρουν ε, τι ε, ε, είναι οι συνέπειες της μεταφοράς της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Οδηγίας προκειμένου και τι έχουν φορτώσει από πάνω τα κράτη-μέλη ε, ως επιπλέον βάρος. Και το τελευταίο, 8, εγώ το έχω ονομάσει ε, καλύτερο έλεγχο ή ελάφρυνση της γραφειοκρατίας. Βέβαια δεν αναφέρεται ρητά αυτό στη συμφωνία. Τι καταφέραμε και τι επιτύχαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε αιτήσια βάση ε, πέρα από την έρευνα που κάνει για την ανάπτυξη και δεν συμμετέχουμε εμείς, θα αναλύει και το γραφειοκρατικό κόστος, δηλαδή κόστος και ωφέλεια ενός ε, νόμου ή μιας ρύθμισης και αυτό θα συνδέεται με ε, το λεγόμενο πρόγραμμα ε, REFIT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο της νομοθεσίας και όπου γίνεται, ε, εφόσον γίνεται, δεν είναι πάντα δυνατό αυτό, θα επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι οικονομίες μπορούν να γίνουν μέσω της ελάφρυσης αυτής της γραφειοκρατίας για να υπάρχει και μάλιστα μετρήσιμο στόχος και σε ορισμένους τομείς να ορίζεται και σε ένα στόχος. Και αυτό μάλλον θα είναι μια νέα υποχρέωση. Βέβαια αυτό είναι μια μάχη που γίνεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σου λέει θες να μειώσεις το διοικητικό άχθος, αλλά δημιουργείς περισσότερο φόρτο σε εμά τώρα, γιατί μας ε, ε, υποχρεώνεις να κάνουμε ετήσια έρευνα για το διοικητικό άκτος. Τώρα βέβαια αυτό είναι η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα αλλά καλό είναι, πάρα πολύ χρήσιμο κάθε χρόνο να έχουμε αυτή την έρευνα. Ωραία, λοιπόν, είναι αυτά, δεν είναι όλα τέλεια. Στη Νέα Διοργανική Συμφωνία συμφωνώ απολύτως με ορισμένα σχόλια που ειδικοί κυκλοφόρησαν. Ε, not to, ε, θα πρέπει όμως να διατηρήσουμε μια ισορροπία. Διαφέρουμε κάπως ε, σχέση εμείς, ε, ε, εμείς διαφέρουμε από το Συμβούλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα μπορούσε να υποστηριχθεί από το Κοινοβούλιο αυτή η συμφωνία νομίζω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Για να δούμε τον κατάλογο των ομιλητών. Κόρμπετ, Πίπερ, Κάουφμαν, Σάιερ, Λεμπρετών και Γκούτελαν. Και μετά οι υπόλοιποι, εντάξει, εντάξει. Ο Ρίτσαρτ πρώτο. σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ και για την παρουσίασή σου. Όπως ξέρεις η ομάδα μου ανησυχούσε και προηγουμένως για αυτή τη συμφωνία και ανησυχούσε ιδιαίτερα μήπως καταλήγαμε σε κάποιο σε ένα ακόμα νεοφιλελεύθερο συμβιβασμό αλλά είδαμε χθες το βράδυ στην ομάδα τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης τη βρίσκουμε αποδεκτή έχει ακόμη σημειώνει και μερικές προόδους και αυτό οφείλεται στην πολύ προσεκτική και λεπτομερή εντολή που έλαβες και την, την ε, συνέταξε μεταξύ άλλων και η ομάδα μου αλλά ίσως και στις διαπραγματευτικές σου ικανότητες και της ομάδας σου. Με αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, να έχουν γίνει μερικές πρόοδοι στον προγραμματισμό, στις κατεξουσιοδότησεις πράξη στη μεταφορά και αποτίμηση της νομοθεσίας εθνικά, την δέουσα διαφάνεια, ακόμα πρέπει αυτό να βελτιωθεί βέβαια, προστατεύει τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων από παρεμβάσεις και επιτρέπει την επιχρήσωση gold plating γιατί τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να εφαρμόσουν ανώτερα υψηλότερα πρότυπα. Αλλά όταν το κάνουν να είναι γνωστό αυτό για να τα βλέπει ο κόσμος καθαρά. Πολλά καλά όλα αυτά. Κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εμάς στην ομάδα μας όπως ξέρεις είναι τι θα γίνει με τις αξιολογήσεις ή τις μελέτες αντικτύπου. Και είχαν τεθεί ορισμένοι όροι πρώτον να είναι απλώς κατευθυντήρες γραμμές και οι πολιτικές αρχές με δημοκρατικές διαδικασίες να παίρνουν τις τελικές αποφάσεις. Το λέει το κείμενο. Είχαμε πει επίσης ότι πρέπει οι μελέτες αυτές να εξετάζουν και το κόστος που θα αντιπροσώπευε η μη εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας ή όπως λέγαμε παλαιότερα της μη Ευρώπης. Να μην λένε δηλαδή μόνο, να μην μιλάνε μόνο για άχθη και βάρη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στο γενικότερο περιβάλλον επιχειρησιακό προστασίας των καταναλωτών και μας το έβαλες και αυτό. Απαλλαγήκαμε επιτέλους από την ιδέα ότι οι αξιολογήσεις γίνονται στο τέλος της διαδικασίας γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι μια τακτική καθυστέρηση αλλά στην αρχή και πλήρως από την Κομισιόν τώρα θα γίνονται για να καταλάβουμε και εμείς πού χρειάζεται να κάνει το Κοινοβούλιο μια μελέτη αντικτύπου. Πρέπει τις λεπτομέρειες να τις ε, καθορίσουμε βέβαια, αλλά όλα αυτά καλά είναι. Και η συμφωνία αυτή είναι αποδεκτή και όπως κάνουμε συνήθως με συνθήκες και τέτοιες συμφωνίες, τι κάνει το Κοινοβούλιο. Εξετάζει και βλέπει αν μπορεί σαν λάστιχο να την επεκτείνει όσο μπορεί, να την τραβήξει στα όρια για να την βελτιώσει. Βέβαια άμα την παρατραβήξει μπορεί και να σπάσει, αλλά υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης των πραγμάτων στον τρόπο εφαρμογής ιδιαίτερα. Η ομάδα μας λοιπόν ικανοποιήθηκε με αυτό το αποτέλεσμα και το εγκρίνει. Αλλά πρέπει να προσθέσω κάτι. Ένας πρωθυπουργός κάποιου κράτους μέλους που δεν θυμάμαι ποιος <laughs> θέλει να μεταρρυθμίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και πηγαίνει στις συνεδριάσεις λέγοντας έχω τέσσερα κυρία θέματα για μεταρρύθμιση. Ίσως Ξέρεις και εσύ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασταμάτητα μεταρρυθμιστική. Συνεχώς μεταρρυθμίζει πολιτική διαδικασίες. Αυτό κάνουμε εβδομάδα την εβδομάδα και μήνα το μήνα. Και είναι και αυτό ένα παράδειγμα τέτοιας αέναης μεταρρύθμισης. Είμαι βέβαιος ότι όλοι εδώ θα χαίρονταν εάν μπορούσαν να πούν σαν την τηλεοπτική σειρά Yes Prime Minister πολύ ωραία είναι ικανή και η Αγγλία να καταρρυθμίσει εάν συμφωνήσουν όλοι ευχαριστώ αν συνεργαστούν όλοι ε, μια στιγμή για αυτό το τελευταίο μπορεί να μην υπήρξα απόλυτα σαφής την περασμένη εβδομάδα πήγα και είδα τον Κάμερον και του εξήγησα τη διαθεσμική και τη, του άρεσε Άρα συμφωνεί και αυτός. Α, τότε θα ξανασκεφτούμε τη θέση μας εμείς. <laughs> Γι' αυτό το είπα αφού εκφράστηκες. Α. Τελειώσατε. Έχουμε ακόμα 8 μιλητές και πρέπει να φύγει ο Γκίστης και μισή. Ναι, ναι, έχω ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι να... Δύο λεπτά ο καθένας ο Μάρκος Πίπα και μετά κάποιος από την ΑΦΚΟ και μετά λοιπόν Μάρκος Πίπα. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος του ΕΛΚ ε, είχα την ευκαιρία και από τη Σκοπιά των Μικρομεσαίων να το συζητήσω με τον Κίφερ Χόφστατ και μερικά σημεία είναι όντως θετικά ας πούμε η ίδια μελέτη αντικτύπου που μπορεί να κάνει τώρα το Κοινοβούλιο, η πλαισίωση του Κοινοβουλίου στις κατεξοδότηση πράξης, το gold plating, όλα αυτά έχουν βελτιωθεί. Υπάρχουν όμως και άλλα. Ωστόσο, πολλοί από εμά στο ΕΛΚ είμαστε απογοητευμένοι. Σε ό,τι αφορά την ε, μεταχείριση ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχει μια παλιά συμφωνία και στην προηγούμενη λέγαμε ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος για τον αντίκτυπο που θα έχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το έχουμε ξαναπεί στον ΚΙ ε, βέβαια το λέει η συμφωνία αλλά το λέει με τελείως αποδυναμωμένο τρόπο και αυτό μας ε, έχει απογοητεύσει βαθύτατα δεύτερον το Συμβούλιο Ελέγχου, αυτό το Scrutiny Board, δεν είναι τόσο ανεξάρτητο όσο θα υφημούσαν ορισμένοι, γιατί είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και οι τρεις εξωτερικοί εμπειρογνώμονες είναι φιλοσικείς ουσιαστικά. Και η διαιτητική λειτουργία που θα είχε το πάνελ το ανεξάρτητο μετά από θυμία από ό,τι ακούω του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εξαιρέθηκε, δηλαδή η ταχεία διαδικασία. Αυτό δεν το κατανοούμε απολύτως. Νομίζουμε ότι ε, τα ε, μειονεκτήματα υπερτερούν των πλεονεκτημάτων και μείναμε στα μισά του δρόμου. Και τέλος, γιατί έγιναν κρυπτό και παραβίστο αυτές οι διαπραγματεύσεις. Εμείς λέμε να έχουμε περισσότερη διαφάνεια. Αυτό θέλουμε να είναι το αποτέλεσμα. Αλλά διαπραγματεύσεις πιο μυστικά πεθαίνεις. Είναι σάτυρα αυτό, είναι φάρσα αυτό που έγινε. Μετά από κάποιες συστάσεις Προέδρου πολιτικής ομάδας, με ένα εισηγητή που ορίστηκε στην αρχή ήταν ο Σούλτς, αυτός έδωσε τη σκητάλη στον επόμενο που ήσασταν εσύ με μηδενική γραπτή ενημέρωση, μηδενική, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και τώρα έρχεσαι ε, μας φαίνεται ένα αποτέλεσμα και το δεχόμαστε ή το απορρίπτουμε. Ε, αυτά τελικά είναι κάτω από τη βάση ως αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Μπορώ να απαντήσω, ο κύριος Φεχόφστατ. Ναι, να απαντήσω ε, αμέσως. Προτιμώ, γιατί δεν θέλω να πλανώνται διάφορε στο ε, αέρα. Πρώτο για τις μικρομεσαίες κύριε Πίπε. Είναι σαφέστατο ότι στη μελέτη αντικτύπου αυτό είναι υποχρεωτικό, είναι δεσμευτικό. Δεν υπάρχει, δεν νοείται μελέτη αντικτύπου χωρί να μελετάμε τον αντίκτυπο στι μικρομεσαίε. Δεν είναι καθόλου εθελούσιο. Το λέει ξεκάθαρα το, το κείμενο. Περιβαλλοντικό, οικονομικό κτλ. αντίκτυπο κυρίω των μικρομεσαίων παντού. Δεύτερον, κάτι απαντάει ο κύριο Πίπερ εκτό μικροφώνου δεν ακούμε. Δεν λέει if possible στο βαθμό του δυνατού, καθόλου δυνατού. Για άλλο θέμα το λέει αυτό και σε άλλη θέση, άλλη παράγραφο του κειμένου. Δεύτερον, μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης για τη μείωση του άχθους και ε, ε, τον έλεγχο και πάλι είναι υποχρεωτικό. Και προβλέπεται τη μείωση του βάρους για τις μικρομεσαίες και κατά την άποψη μου αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε ένα ωραίο κείμενο που να είναι δεσμευτικό για τις μικρομεσαίες, όχι και στα δύο, και στο αντίκτυπο και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Το έχουμε προβλέψει κυρίως για τις μικρομεσαίες. Το πρώτο αυτό. Δεύτερον, φερστέκ τίποτε κρυπτό και μυστικά. Στη γλώσσα μου αυτό σημαίνει ότι κάναμε μυστικές διαπραγματεύσεις. Αν ήταν αυτές μυστικές διαπραγματεύσεις, Ήταν ασάνοιχτες οι πόρτες, οι μυστικέ. Κάθε φορά, μετά από κάθε γύρο, πήγαινα στη διάσκεψη των Προέδρων, παρουσία του Προέδρου της Γιούρη και ε, της Προέδρου της ΑΦΚΟ για να κάνουμε την ενημέρωση κάθε φορά, το debriefing. Και έχω δει σχεδόν όλες τις ομάδες εργασίας όλων των πολιτικών ομάδων και στο ΕΛΚ και στους σοσιαλιστές και δημοκράτες όχι ακριβώς, αλλά τουλάχιστον με τον πρόεδρο της ομάδας εργασίας, τον κύριο Κόρμπετ Έχω ε, κάνει συνεδριάσεις με τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές και με τους πρασίνους και πού δεν πήγα, ακόμα και στην EFTD ένα τμήμα τους, γιατί έχετε και εκεί δύο συνιστώσεις. Δύο μεγάλες εθνικές αντιπροσωπίες. Δεν είναι ουσιαστικά ομάδα, μια τεχνική φόρμουλα έχουν βρει και τα έχουν ενώσει. Ε, ναι, μου είχαν ζητήσει οι πράσινοι και η ΕΝΕΦ είχα πάει και σε αυτούς. Και τρεις συνεδριάσεις είχα μαζί σας και μία μόνο με τον κύριο Κόρμπετ. Μπορώ να σας τα πω αυτά ξεκάθαρα. Κύριε Κόρμπετ, σας έριξε ο κύριος ε, Πίπερ και σας έχει κερδίσει. Και μετά έρχεται και μου λέτε ότι είναι μυστικές οι διαπραγματεύσεις. Εγώ ξέρω κάτι άλλες μυστικές διαπραγματεύσεις. Ως Πρωθυπουργός ε, σε έχω κάνει και αυτές πολλές φορές τελείως. Καμία σχέση δεν έχει με τις παρουσίες για τη διοργανική συμφωνία. Ευχαριστώ, ο Τζότς Σόπφιν. Thank you, Uh, Τρεις ερωτήσεις. Το ανεξάρτητο Συμβούλιο Αξιολόγησης Αντικτύπου. Ε, ποια ακριβώς θα είναι, τι διαφάνεια θα έχει, ε, μπορεί κανείς να εφεσιβάλει τα αποτελέσματα, τα πορίσματα κλπ. Περισσότερες λεπτομέρειες λοιπόν. Δεύτερο ερώτημα. Όταν το Συμβούλιο αυτό θα αναλαβεί δράση ε, θα περιλαμβάνονται ε, ρήτρες ε, αποτυχίας, sunset, ρήτρες κατάληξης, εκπνοής κλπ. Τρίτον, θα γίνει μια συγκριτική αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών, θα υφίσταται κάποιος μηχανισμός ώστε να ενθαρρύνονται τα κράτη-μέλη να αφαιρούν το gold plating αν είναι υπερβολικά πολύ. Uh, uh, Είπα ότι έστειλα την επιστολή του κυρίου Τίμερμανς ε, με τρεις σελίδες λεπτομέρειες. Είναι αυτές ακριβώς οι οποίες, τις οποίες ε, ε, ζητάτε. Το έστειλα και στις δύο επιτροπές. Από ό,τι φαίνεται δεν τις έχετε πάρει, αλλά κάποιοι εδώ αριστερά και δεξιά κρατούν αυτή την επιστολή στα χέρια τους οπότε θα ήθελα να γίνουν αντίγραφα για να μοιραστούν. Ακριβώς διότι και εγώ ζήτησα τα ίδια ακριβώς πράγματα από τον κύριο Τίμερμας και μου απάντησε μέσω αυτής της επιστολής. Έχει ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου. Δυστυχώς όμως από ό,τι φαίνεται δεν έχει αποσταλεί σε όλους. Θα μπορούσατε λοιπόν να, κάνετε, να κάνουν οι υπηρεσίε μα ένα αντίγραφο και να διανεμηθεί. Για να δείτε και τι λεπτομέρειε, να μου πείτε αν αρκετέ ή όχι. Ευχαριστώ. Το, για το gold plating ε, δεν ξέρω αν έχετε κάποια απάντηση. Ποια ήταν η ερώτησή σας? Να σας την ξαναπώ θα γίνει μια συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών. Δηλαδή θα υφίσταται μηχανισμός ε, που να λέει το πώς θα πρέπει να γίνεται η εφαρμογή και να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αφαιρούν τον gold plating. Όχι. Η απάντηση είναι ρητά όχι. Για τον εξή απλό λόγο. Διότι δεν απαγορεύεται το gold plating. αν κατά τη μεταγραφή μιας οδηγίας ε, ε μέσω νομοθεσίας ή μέσω ε, διατάγματος, ε, υπουργικού διατάγματος ας πούμε, τι γίνεται. Μεταγράφεται την οδηγία, χρειάστηκε να το εξηγήσω αυτό και στη διαπραγμάτευση, γιατί όλοι μιλούσαν για gold plating, αλλά κανένα δεν είχε κάνει gold plating. Οπότε τους είπα, σας εξηγήσω πώς λειτουργεί, εγώ που ξέρω. Έχουμε το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να μεταγράψει μια οδηγία. Και πολλοί έχουν διάφορες πολύ ωραίες ιδέες και λένε κάποιοι υπουργοί. Μια και θα μεταγράψουμε την οδηγία αυτή, δεν μπορούμε στο, στην ίδια νομοθετική πράξη, στο ίδιο διάταγμα να προσθέσουμε και αυτό. Γιατί μου χρειάζεται, λέει ο κάθε υπουργό. Αντί να το κάνουμε χωριστά, ας χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη νομοθετική πράξη, νομοσχέδιο κλπ. Ε, για να προσθέσουμε και κάποιες άλλες διατάξεις. Οπότε, πολύ συχνά ε, σε κάποιο νομοσχέδιο ε, έχουμε και μια, ένα τελευταίο κεφάλαιο με διάφορες διατάξεις. Έτσι ονομάζεται, έτσι είναι ο τίτλος συνήθως όπου προστίθενται διάφορα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση ή μόνο ακροθυγώς σχετίζονται με το, με το ίδιο το νομοσχέδιο. Δεν θέλουμε να το απαγορεύσουμε, δεν θα μπορούσαμε να το απαγορεύσουμε. Το μόνο που ήταν δυνατό να γίνει είναι ότι όταν γίνεται gold plating θα πρέπει να αναφέρεται ρητά και ότι η Κομισιόν θα παρακολουθεί πλέον το gold plating και θα το δημοσιεύει θα λέει αυτό το κομμάτι αφορά την μεταγραφή, εκείνο το κομμάτι δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και είναι προσθήκες σε εθνικό επίπεδο. Όχι, δεν θα έχουμε όμως ε, συγκριτική αξιολόγηση, βέλτιση των πρακτικών κλπ. κλπ. Ε, δεν θα... Ε, οι, οι, οι Βρετανοί ας πούμε τι κάνουνε, μεταγράφουν την οδηγία λέξη προς λέξη. Και οποιασδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνουν γίνονται ξεχωριστά σε ένα άλλο νομοθετικό κείμενο. Ε, ε αυτή η μέθοδος είναι διαφορετική, πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες χώρες. Ε, σε άλλες χώρες η ε, μεταγραφή χρησιμοποιείται και τυχαίνει κατάχρηση πολλές φορές. Ε, είναι πολύ συχνά θύμα των συγκρούσεων μεταξύ συμμάχων, κυβερνητικών συμμάχων. Κύριε Κάουφμαν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σας κύριος, κύριε Φερχόφστα, εσένα Γκή. Πρέπει να πω ότι με έκπληξη έμαθα ότι ολοκληρώθηκε η συμφωνία πριν τα τέλη του έτους. Την τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί στη νομική επιτροπή δεν συμμεριζόμουν αυτή την αισιοδοξία, αλλά τόσο το καλύτερο. Δεύτερον, ε, συμφωνώ απολύτως ε, με αυτό που είπε ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ για την ομάδα μας, ότι είναι καλό το κείμενο και θα ήταν πάρα πολύ καλό να το εγκρίνει συνολικά το Κοινοβούλιο. Είναι πολλά τα θετικά, τα οποία ήδη αναφέρθηκαν. Εγώ θέλω να μιλήσω μόνο για τη μελέτη αντικτύπου στη δική μου έκθεση που δυστυχώς δεν έχει φτάσει στην Ολομέλεια. Ακριβώς αυτή τη γραμμή υπερασπιστήκαμε για τη μελέτη αντικτύπου και είναι πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω για τα τρία θεσμικά όργανα να προχωρήσουμε τον τρόπο που περιέγραψες και που συμφώνησαν. Βέβαια τίποτα δεν είναι τέλειο στο μάταιο του το κόσμο. Αλλά στην παράγραφο 14 γίνεται ε, λόγος για δημόσια διαβούλευση και διαβούλευση των ενεχομένων. Βέβαια αυτό αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι δεν είναι. Αλλά αν δεν αφαίρεται πουθενά η διαβούλευση της κοινωνίας των πολιτών, η κοινωνία των πολιτών, απλώς γίνεται λόγος για μικρομεσαίες και άλλους τελικούς χρήστες. Αυτό μου φαίνεται μάλλον ομολογία αποτυχίας. Δεν ξέρω μήπως θα χρειαστεί να συνεχιστεί αυτός ο καυγάς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ένα τελευταίο, το θέμα των τριμερών διαλόγων. Επίσης χαίρομαι που υπάρχει μια μικρή ρήτρα ε, που ανοίγει ε, λίγο ε, μια πόρτα. Πώς θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια πέρα από αυτό που είπες για την Grand Place που συμφωνώ αλλά υπάρχουν κανόνες τους οποίους δεν εφαρμόζουμε από ό,τι φαίνεται ε, με ακρίβεια για τους τριμερείς διαλόγους, ούτε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο δηλαδή. Καλούμεθα όλοι να δράσουμε και ελπίζω οι ε, συνομιλίες να καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα αποδεκτό για όλους και κατανοητό για τους πολίτες. Τι θέλουμε να κάνουμε στην νομοθεσία. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Για τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους ζήτησαν οι δύο επιτροπές να γίνει αυτή η διαβούλευση μετά την έγκριση. Αυτό βέβαια βγήκε από το κείμενο. be very careful. Αλλά να είμαστε προσεκτικοί. Σβήστηκε, αλλά μπορεί παρόλα αυτά να γίνει. Α, κομισιόν. Εγώ το βρίσκω πολύ λανθασμένη ιδέα ενώ αρχίζει μια νομοθετική διαδικασία ταυτόχρονα να αρχίζει η διαβούλευση ενδιαφερομένων γιατί έτσι οργανώνονται τα lobbying άκου λέει την ίδια στιγμή έτσι απλώς παρεμβαίνει μια διαδικασία στην άλλη δεν το δεχόμαστε ούτε το Συμβούλιο γι' αυτό σβήστηκε από το κείμενο και εγώ λέω κάτι πολύ απλό εάν ξανά θελήσουν να κάνουν μετά την έγκριση από το από το κολέγιο την ε, διαβούλευση των ενδιαφερομένων να το κάνουν γνωρίζοντας ότι παίρνουν πολύ μεγάλο, αναλαμβάνουν πολύ μεγάλο κίνδυνο. Αυτό ε, αυτό πιστεύω εγώ, αυτό πιστεύω. Επιβραδύνουν την νομοθετική διαδικασία. Εμείς και το Συμβούλιο το σβήσαμε. Αν θέλουν όμως να επανέλθουν και που «Α, να, χρειαζόμαστε πέντε εβδομάδες και τέτοια». Για μένα είναι απλό. Τότε η νομοθετική διαδικασία θα αρχίσει από το Κοινοβούλιο αυτές τις 5-8 εβδομάδες μετά. Εγώ ποτέ δεν θα δεχτώ παράλληλα τα δύο πράγματα. Ποτέ! Γιατί έτσι υπονομεύεται η νομοθετική διαδικασία. Δεν πρέπει να οργανώνονται τα λόμπι την ίδια στιγμή που και εμεί κάνουμε την νομοθετική μα εξέταση. Τέλο πάντων, έχει σβήσει από το, έχει από το κείμενο. Αλλά να το προσέχουμε. Μήπως επανέλθει από την πίσω πόρτα. Αυτή η ανόητη ιδέα. Ευχαριστώ. Μπαν πάνε μας δώσει. Ε, τι να κάνεις. ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σου. Ε, συμφωνώ με την κατεύθυνση του εγγράφου. Έχουμε μια καινούργια διαδικασία ε, που θα μας βοηθήσει πολύ. Έλεγα λοιπόν που ότι θέλω να σε ευχαριστήσω για τη δουλειά σου. Θεωρώ ότι πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την μείωση του διοικητικού άχθους. Θα ήθελα να έχει προβληθεί και καλύτερη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ιδιαίτερα στην αρχή της εκ των υστέρων ανάλυσης δηλαδή της ανάλυσης μετά την εφαρμογή της συμφωνίας. Το άρθρο 23 είναι απλώς δηλωτικό. Ε, λέει ότι θα ενημερώνονται τα εθνικά κοινοβούλια καλύτερα σε καθένα από τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας. Αυτό συμπεριλαμβάνεται. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να, θα πρέπει να θεωρείται ως εταίρος των Εθνικών Κοινοβουλίων και να βελτιωθεί η συνολικά διαδικασία ενημερωσή του. Ο κ. τα αναφέρεται σε πολλά σημεία του εγγράφου, αλλά σίγουρα αυτό που δεν κάναμε ε, και δεν μπορεί να γίνει είναι ε, να αλλάξουμε την θεσμική ισορροπία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια όπως έχει καταγραφεί στην ε, συνθήκη ε, η, δεν είναι δυνατόν με μια διοργανική συμφωνία ή μέσω νόμου να αλλάξουν οι συνθήκες. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται να δίνουμε περισσότερο βάρος στα Εθνικά Κοινοβούλια σε ό,τι αφορά την εξέταση των νομοθετικών κειμένων κλπ. Αλλά όλα αυτά προβλέπονται στη συνθήκη. Μπορούμε να επικρίνουμε τη συνθήκη. Κάποιοι ε, λένε ότι Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων κλπ. Αλλά ε, δεν είναι τη στιγμή σε αυτή η συζήτηση. Ε, η ΑΦΚΟ ετοιμάζει δύο εκθέσεις για τη θεσμική δομή εντός των συνθήκων, στο πλαίσιο συνθήκων και την μελλοντική θεσμική δομή. Εκεί μπορούμε να τα συζητήσουμε αλλά δεν ήταν δυνατόν όλα αυτά να συζητηθούν στο πλαίσιο μιας, της διαπραγμάτευσης μιας ε, διοργανικής ε, ε, συμφωνίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ισορροπία μεταξύ του ρόλου των θεσμικών οργάνων ή των κοινοβουλίων. well, thank you very much and thank you for your work and um, I would say that um, especially in uh, area of uh, delegated... Ευχαριστώ πολύ ιδιαίτερα για τις κατεξοδότητες και τις πράξεις. Στην Επιτροπή μας ε, ε, έχουμε κάνει παρουσιάσεις και κατηδίαν τα είπαμε. Βεβαίως πολύ σκληρή δουλειά και φαίνεται. Η συνθήκη της Λισαβόνας δημιούργησε μια ιδιάζουσα κατάσταση εδώ. Γιατί ε, δύο ισότιμα μέρη θα πρέπει να αγωνίζονται για το ίδιο πράγμα και το θέμα είναι πώς τα διαθετείς αυτά. Δηλαδή, αν βάλεις μια σοκολάτα... Ε, στη μέση του δωματίου και είναι δύο παιδιά και έχουν ίσο δικαίωμα, θα χυμίξουν να την πάρουν. Και ανάλογα με το χρώμα της σοκολάτας, το ένα παιδί έχει περισσότερα δικαιώματα και το άλλο λιγότερα. Ε, δηλαδή δεν είναι ε, πολύ, ε, ακριβώς η αντιστοίχηση και η ισότητα Κοινοβουλίου Συμφουλίου. Ε, χαίρομαι και εκτιμώ για την απόπειρα που κάνετε για να συμμετέχουμε και στις εθνικές διαβουλεύσεις ενώ με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες και η σχετική διαβούλευση ήταν κάτι ε, ε, που ε, ήταν μια μάχη που δώσαμε και μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν παραδοθήκαμε. Έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά συμφωνώ ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένω να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, αν θέλουν τόσο πολύ αυτή τη σοκολάτα, τους δώσουμε ένα κομματάκι και μετά συνεχίζουμε. Ε, ορισμός υπάρχει σύμφωνα με τον οποίο χαρακτηρίζουμε ένα πράγμα ζάχαρη ή σοκολάτα, αλλά το απέναντι μέρος δεν τα δέχεται όλα αυτά. Ε, ε, ε, λοιπόν, θα προτιμούσα να έχουμε κάποιο είδους κοινά κριτήρια. Ιδιαίτερα για την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων που είναι αρμόδια για την οριζόντια εκτέλεση στο Κοινοβούλιο πώς θα γίνεται η διάκριση ανάμεσα στη κατεξοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις, κάνει ε, εκθέσεις, παρακολούθησης κτλ. Και η διάσκεψη των Προέδρων το έχει εξετάσει και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Και ίσως η ζωή μας είναι λίγο πιο εύκολη αργότερα. Θα επανέλθω όμως για να το ελέγξω, αν πραγματικά είναι ευκολός. Γιατί είναι πολύ μεγάλη η υποχώρηση και η παραχώρηση που κάνουμε στο Συμβούλιο εδώ και θα πρέπει να επαγρυπνούμε ε, και να διαφυλάξουμε τις δικές μας αρμοδιότητες και εξουσίες. Τώρα δεν έχουμε καμία εξουσία γιατί δεν έχουν κινηθεί καθόλου τα πράγματα και θα μπορούσαν τελικά να μπλοκάρουν όλη την νομοθετική διαδικασία αν δεν αντιδράσουμε. Ε, θα πρέπει να επιδείξει την ίδια ε, καλή προαίρεση και το Συμβούλιο. Λοιπόν, ας το κάνουμε. Αυτό πείραμα είναι. Ναι. Καλή είναι η ιδέα. Ε, είναι καλό αυτό να γίνει αυτή η συζήτηση για το διαχωρισμό, να δούμε ποια πράξη θα είναι τι και να το εκτιμήσουμε εκ των υστέρων, να αξιολογήσουμε πώς θα έχει λειτουργήσει. Ε, συμφωνώ πολύ τους κύριε Σάγερ. Ο κύριος Χρυσόγωνος, παρακαλώ. Thank you. Uh, we have discussed the, the outcome. Συζητήσαμε το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων χτες στην ΚΟΕ και μπορώ να πω ότι είμαστε αρκετά διστακτικοί. Πρώτον, σε φορά την διαφάνεια. Ε, υπάρχει μια γενικόλογη διατύπωση για την ανάγκη μεγαλύτερη διαφάνεια στην νομοθετική διαδικασία, αλλά βλέπουμε λίγες απτές ε, δεσμεύσεις ε, σε ό,τι αφορά τις κυβερνήσεις και το κοινό. Σε ό,τι αφορά τη μελέτη, τις μελέτες αντικτύπου, η συμπερίληψη ε, των, της κοινωνικής στοιχής και της πραγματικής τυχή είναι κάτι θετικό, αλλά οι επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, έχουν την προτεραιότητα στις ε, μελέτες αυτές ή στις εκ των υστέρων αξιολογήσεις ή Επιπλέον, δεν αναφέρονται ρητά τα συνδικάτα. Το συμπεράσμα μας γενικότερα είναι ότι ε, πέραν του ενισχυμένου ρόλου στον πολιτικό ετήσιο προγραμματισμό, ο ρόλος του Κοινοβουλίου δεν ενισχύεται σημαντικά από αυτή τη Οργανική Συμφωνία. Αντιθέτως, ε, το refit ε, ενισχύεται με αναφορές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και με τη ε, συνεχείς αναφορές στο διοικητικό άκθος. τέλος, η εισαγωγή αυτού του Συμβουλίου Αξιολόγησης Εμπειρογνώμων για την αξιολόγηση μπορεί να μειώσει το ρόλο του Κοινοβουλίου. Και τι θα γίνει αν η πρόταση λάβει μια αρνητική αξιολόγηση. Παρόλο ότι μιλούμε για καλύτερη νομοθέτηση, ο στόχος τελικά είναι η ε, απελευθέρωση και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την συμφωνία. Ε, χαίρομαι διότι ε, ε, πείθετε τον κύριο Πίπερ για τα επιχείρηματά μου. Ε, ήταν πολύ αντικειμενική η τοποθέτησή σας εκτός του του ΕΛΚ. Ήταν πολύ αντικειμενική. Και, και εκτός της Άλντε. Ευχαριστώ κύριο Λεβρετό. Ζητώ συγγνώμη Κύριε Φερχόφστατ, πάντα με χαρά σας ακούω, ακόμα και αν δεν συμφωνώ ε, κατά ανάγκη μαζί σας. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την υπερβολική ρύθμιση και νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπαίνει σε μια ομοσπονδιακή διαδικασία που επιταχύνεται, ενώ ο κόσμος απομακρύνεται, περίεργο φαινόμενο. 80% των εθνικών νόμων δεν είναι παρά η μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών. Τα εθνικά κοινοβούλια έχουν μόνο περιθωριακή, περιθωριακή νομοθετική εξουσία, πόσο μάλλον που η αρχή της επικουρικότητας παραβιάζεται. Σε αυτή την ε, προοπτική λοιπόν της υπερβολικής ρύθμισης πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λένε. Ότι ένα κράτος θα πρέπει να δηλώνει τι ε, επιπλέον εγκρίνει όταν μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι ανακατεύεται ξανά η Ευρωπαϊκή Ένωση στην νομοθετική ε, δραστηριότητα και εξουσία των κρατών μελών που είναι ήδη περιφερειακή και περιθωριακή. Ήδη κατέχει το 80% η Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα διεισδύει ε, και στο υπόλοιπο 20%. Και πάλι φθηνά τη γλιτώσαμε γιατί η Κομισιόν ήθελε να το πάει ακόμα παραπέρα. Και εσείς κύριε Φερχόφστατ θέλετε να ε, απαγορεύσετε την υπερβολική ρύθμιση. Ε, στο όνομα λοιπόν της κυριαρχίας των κρατών μελών εγώ τα καταδικάζω όλα αυτά και εξ ονόματος της ομάδας μου δεν θέλω τα εθνικά κοινοβούλια, πόσο μάλλον η Γαλλική Εθνική Συνέλευση θα γίνουν ε, θέατρα σκιών. Μα αυτό το 85% λέει ο κύριος Φερχόφστατ δεν είναι 85% γιατί θα φανεί ότι είναι πολύ λιγότερο. Αλλά το 85% είναι ένα ε, νούμερο που προκύπτει από το επιχρήσωμα του gold plating των κρατών μελών. Που με για τους με χαρά τους. Εγώ δεν απαγορεύω τίποτα. Το κείμενο το απαγορεύει. Ε, ε ο κανονισμός, ε, νομοθετικά κείμενα, ε, τα διατάγματα βασιλικά ή ε, υπουργικά. Δεν είναι 85%, είναι λιγότερο. Μπορεί να μην σας αρέσει γιατί δεν σας βοηθάει στην πολιτική σας μάχη, αλλά δουλειά μας δεν είναι να σας βοηθάμε εσά στην πολιτική σας μάχη. Το αντίθετο, για να σας καταπολεμούμε και να αντιπαλεύουμε. Thank you and the last... Ευχαριστώ. Η κυρία τελευταία. Thank you, and uh, Thank Σας ευχαριστώ για τη σκληρή σας δουλειά. Είναι και ήταν και ο συνάδελφος εδώ που είπε μερικά πράγματα που δεν θα επαναλάβω, αλλά θα ήθελα να τονίσω μόνο το γεγονός ότι για το άχθος, το άχθος αναφέρεται 11 φορές στο κείμενο. Άχθος και δεν κατάλαβα ποιες είναι οι θετικές επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και γιατί έχει λέει μεγαλύτερες επιπτώσεις πιο θετικές από ό,τι η Εθνική Νομοθεσία. Ούτε συμφωνώ ότι πρέπει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να μην τη βλέπουμε σαν ευκαιρία αλλά σαν άχθος, έτσι λέει. Ούτε αποκλεί ποσοτικού στόχους για τη μείωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αυτό νομίζω ότι δεν είναι σωστό, είναι αντιπαραγωγικό που λένε. Επίσης νομίζω ότι πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία και να υπάρξει απλοποίηση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Χωρίς όμως αυτό να μας αποπροσανατολίζει από τους στόχους μας. Οι στόχοι αυτοί καθορίζονται από τις συνθήκες. Αλλά δεν βρίσκονται στην καρδιά του κειμένου αυτού. Αντί να τονίζει τα κυριότερα προβλήματα της Ένωσης, η βασική του αρχή είναι thinking small. Εγώ δέχομαι τη σημασία της προώθησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να παίξουν ρόλο, να συμμετάσχουν. Είναι το κλειδί για την επιτυχία της Ένωσης. Τέλος δε, η Ένωση αντιμετωπίζει τώρα τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι τώρα. πυλές τρομοκρατίες, κλιματολογικές αλλαγές, οι πρόσφυγες, εκκλήσεις για κλείσιμο των συνόρων, αυξημένη έλεγχη στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία λέγω βλέπουμε ότι θεμελιώδεις ελευθερίες όπως η ελευθερία του λόγου κάνουν επίθεση και γι' αυτό πρέπει να κρατήσουμε την προσοχή μας ζωντανή στα βασικά. Βέβαια πρέπει να γίνει προσπάθεια απλοποίησης αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα είναι αποτελεσμάτικη ε, και θα επιτυγχάνει τους κύριους στόχους της και από τη συνθήκη και από τη στρατηγική του 2020. Μάλλον θα συμφωνείτε με πολλά από αυτά που είπα, αλλά λυπάμαι δεν το βλέπω στο κείμενό σας. Κοιτάξτε για το βασικό που είπατε. Το λέει η συμφωνία ότι σε κάθε αξιολόγηση, το είπε και ο κύριος Κόρμπετ, θα υπάρχει, θα αναφέρεται και το κόστος της μη Ευρώπης. Τι σημαίνει αυτό. Ότι αν είναι χαμηλότερο το διοικητικό άχθος, θα είναι χαμηλότερο το διοικητικό άχθος αν έχουμε μία κοινή νομοθεσία αντί 28 διαφορετικά εθνικά επίπεδα. Αυτό είναι. Το κόστος της μη Ευρώπης είναι αυτό. Σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει εθνική, ε, ενωσιακή νομοθεσία θα συνεχίσουν να υπάρχουν 28 διαφορετικές εθνικές. Και αυτό είναι περισσότερο διοικητικό άχθος. So, uh, uh, reduced administrative burden is is not only, oh, reduce uh, legislation on the European level, it is also... Επομένως, μια ευρωπαϊκή λύση, όποτε μπορεί, θα αντικαθιστά 28 διαφορετικές, διαφορετικά άχουθη γραφειοκρατίες, δυσκολίες σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό το λέει ρητά στο τμήμα αυτό του κειμένου. Το κόστος της μη Ευρώπης, πώς να σας το πω. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση, κύριο Σβόμποντα. Uh, Στη διάσκεψη των Προέδρων έχω συμμετάσχει ε, και με ρώτησαν κάτι και δεν έχω απάντηση. Ποιο είναι το συμφέρον του Κοινοβουλίου να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις πριν τα Χριστούγεννα και να αφήσουμε διάφορα πράγματα ε, στις κατεξοδότηση ε, πράξης και τα λοιπά ημιτελή. Μα όταν αρχίσαμε αυτή τη διαπραγμάτευση για να είμαι πολύ ειλικρινή, στην αρχή ήταν πολύ θετική η αντίδραση της Προεδρίας του Λουξεμβούργου. Και αυτό το εκτιμήσαμε πάρα πολύ. Ο κύριος Νικολά Σμιτ ε, διαπραγματεύτηκε από πλευρά του Συμβούλου και ήταν πάρα πολύ πρόθυμος. Και, είπαμε ότι, θεωρήσαμε ότι πολύ καλύτερο θα ήταν να ολοκληρωθεί με εκείνον. And to παρά να ξανανοίξει το όλο θέμα της διαπραγμάτευσης με τη νέα Προεδρία. Δεν θα πω τίποτα για την Ολλανδική Προεδρία, γιατί έχω φίλους στην κυβέρνηση, σταματώ εδώ. Αλλά, ε, ο νόν, νοήτο. Ε, Μπορείτε να πείτε κι άλλα πριν σας αφήσουμε να φύγετε. Όχι, όχι, ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το πείραμα. Ε, να μην διαπραγματεύουμε ως Συμβούλιο όπως στο παρελθόν, αλλά ως Κοινοβούλιο. Of, of, of the Uh, and, uh... Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία πρέπει να σας πω. Ξέρω ότι ακούσαμε επικρίσεις ότι είναι καλό αυτό το να έχει ένα διαπραγματευτεί από το Κοινοβούλιο ε, με την υποστήριξη της διάσκεψης των Προέδρων της Γιούρη και της ΣΑΦΚΟ. Δεν ήταν κακή η εμπειρία γιατί απέναντι μπορώ να σας πω ότι είχαν ένα διαπραγματευτεί από το Συμβούλιο, έναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν θετική εμπειρία και ελπίζω να έχετε κι εσείς την ίδια αίσθηση όταν ε, διαβάσετε το αποτέλεσμα. Είπα όμως και στον κύριο Σούλτς και στη διάσκεψη των Προέδρων ότι αν θέλετε κάποιον για τις διεθνείς συμφωνίες να ψάξετε αλλού, έτσι, εγώ εδώ έδωκα. Τους είπα. Oui, c'est le voleur qui devient policier. De temps en temps, c'est Εντάξει, καμιά φορά γίνονται και κλέφτες αστυνόμοι. Το αντίθετο όχι. Αστυνόμοι, κλέφτες και αυτό θα έχει πλάκα. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κίφερ Χόφστατ. Ως πρόεδρος της ΑΦΚΟ, σας ζητώ να φύγετε όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί έχουμε συνεδρίες των συντονιστών και διερμηνία μέχρι τις 6. Στο καλό να πάτε οι υπόλοιποι.